Thanks a lot. Ladies and gentlemen, welcome on the uh, evening session. The sitting is... Uh, Επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας και ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της συνέσιας διάταξης. Δήλωση της Κομισιόν για την απόφαση του Ευρωπαϊκού